Okay, everybody, can you take your... Πολύ καλά. Μήπως μπορείτε να καθίσετε. Μου λένε ότι δεν θα αργήσουμε, αλλά αν αργήσουμε, τότε θα δώσω την προεδρία σε άλλον. Βλέπετε εδώ, η ομάδα μου έχει αναπληρωματικούς, δεν έχουμε πολλούς, δεν βλέπουμε κανέναν, λοιπόν. Έχουν όλη την κάρτα τους. Η Αλήν δεν την έχει άλλος. Μπορεί να μην χρειαστούν, αλλά όσοι τις έχουν να τις τοποθετήσουν παρακαλώ. Εσείς θα ψηφίζετε, εγώ όχι, μήπως χρειαστεί να φύγω επιγόντως. Λοιπόν, σχέδιο έκθεσης Αγκόκ για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών κλπ. Α, η Αλήν βρήκε την κάρτα της. υπάρχουν συμβιβασμοί και μερικές αποσύρσεις Λοιπόν. Γκούναρ δεν έχεις κάρτα. Βλέποντας τον κατάλογο ψηφοφορίας υπάρχουν συμβιβασμοί που έγιναν δεκτοί αλλά δεν τους γράφει. Α, πάντων. Ο, με μερικούς συμβιβασμούς τους υποστηρίζει και το έλκα αλλά δεν το γράφει. Θα το λέω κάθε φορά, θα το λέω, μάλιστα να με κοιτάζεις και θα σου κάνουν νοήματα. Μάλιστα. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό το πράγμα εδώ μπροστά μας, είναι μία κάμερα πολλαπλής λήψεως, πολλαπλών κεφαλών. Είναι για τα μέσα, για τα μέσα. Είναι η κοινοβουλευτική υπηρεσία, όχι τίποτα εξωτερικό. Γι' αυτό να χαμογελάτε παρακαλώ, αλλά δεν έχει ήχο, είναι χωρίς ήχο. Λοιπόν, λοιπόν θα ψηφίσουμε. Τροπολογία 50 υπέρ τα και εγκρίθηκε. 51 υπέρ Α, όχι, όχι, καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει. Συμβιβασμός α υπέρ. Κατά, έχεις. Εγκρίνεται. 53 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται αν δεν απατώμε. Αν θέλετε μπορούμε να επαληθεύσουμε, αν θέλετε. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλες και όλοι. Ε, ορίστε κύριε Μπούλμαν γρήγορα σας παρακαλώ. Συντομεύετε. Το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί. Αν και ήδη είναι 28 υπέρ και 2 κατά, οπότε ό,τι και να γίνει λοιπόν. Εγκρίνεται και αυτό. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Α, είναι σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ποιες μου φαίνεται ότι εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά ποιες ε, και αυτό 56 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 57 υπέρ κατά ποιες κρίνεται 58 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται συμβιβαστική β έχει αποσυρθεί 59 ε, με προφορική τοποποίηση των πρασίνων ε, υπέρ Α, καλά. Καλά. Την προφορική θέλετε να ψηφίσουμε χωριστά μόνη της. Την προφορική. Καλά, τότε την προφορική. Έτσι έχουν ζητήσει πρώτα. Αν θα συμπεριληφθεί η προφορική ή όχι. Λοιπόν, συμπεριλαμβάνουμε την προφορική υπέρ της συμπερίληψης της προφορικής. Τα. Τη συμπερίληψης της προφορικής αποχές δεν θα συμπεριληφθεί η προφορική. Θα ψηφίσουμε τώρα το αρχικό της τροπολογίας. 59. Υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική γάμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα έχει αποσυρθεί. Προπολογία 61 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το, ε, η συμβαστική ε έχει αποσυρθεί 62 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.

Είμαστε στην 66 λοιπόν υπέρ. Κατά οχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά οχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται 72 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Δύο, λέει πάλι η πρόεδρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 κατά πίπτη, συμβιβαστική σιγματά, F, δηλαδή, υπέρ, κατά εποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται οι υπόλοιπες καταπίπτουν εδώ μέχρι τον συμβιβασμό ζήτα. Λοιπόν, Συμβιβασμός Ζ έχει αποσυρθεί λοιπόν, άρα η 81 υπέρ. Γκούναρ, δική σου δεν είναι η 81, δική σου είναι λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 84 άρχεται η ψηφοφορία έληξε 21 υπέρ 23 κατά απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 με μια προφορική προσθήκη και μελλοντικέ γενιές 86 λοιπόν με αυτή τη διατύπωση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γνωμοδότηση προϋπόλ παράγραφο 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπόλ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. μήπω μπορούμε όλε τι γνωμοδοτήσεις του προϋπόλ μαζί, όχι. Προϋπόλ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπόλ 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπόλ 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπόλ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές, θα επαληθεύσουμε για την 88. Έληξε. Εγκρίνεται 24 με 19. Οι 89 και 90 καταπίπτουν. 91 υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. Συμβιβαστική ήττα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβιβαστική θήτα υπέρ κατά εποχές ας το επαληθεύσω καλύτερα Ηλεκτρονικά είπαμε, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, νομίζω ψήφισαν όλοι, λίγη η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 22-21. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Χες. Yes. 97 Καταπίπτει 98 όμως δεν καταπίπτει υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 99. Α, όχι, έχει καταπέσει, καταπέσει λόγω του 98. Όχι! Όχι. Μα εδώ γράφει ε, στην 98 αν εγκριθεί 99 καταπίπτει. Έτσι γράφει στον κατάλογο. Δεξιά. Α, ναι, ναι, έχει καταπέσει λοιπόν η 94 και η 100 επίσης λόγω της 96. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και άρα καταπίπτουν όλες οι υπόλοιπες για την 8. 105 έχει αποσυρθεί. 106 υπέρ, κατά, ποιες κρίνεται 107 θα πέσει και η 8. Συμβιβασμός Ι, υπέρ, κατά, ποιες κρίνεται 112 υπέρ, κατά, ποιες κρίνεται συμβιβασμός Ι, α, υπέρ, κατά ποιες κρίνεται συμβιβασμός ΙΒ υπέρ κατά ποιες επαλήθευση για το συμβιβασμό ΙΒ L δηλαδή λατινικό έληξε 19 υπέρ 24 ε, κατά απερίφθη α δεν είχα κάρτα εγώ δεν είχα Έλα να αφού απερίφθη, απερίφθη. Λοιπόν. Και μάλιστα κάρα απερίφθη. Λοιπόν, πάμε τώρα στην 115 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Το ΕΛΚ ήταν κατά. 116. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ τα δεν σηκώνουν όλοι το χέρι 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι υπόλοιπες τις 13 καταπίπτουν προϋπόλ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προϋπόλε 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 της εικόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές να την ξαναδούμε την 122 παρακαλώ. Πήφησαν όλοι. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα γάμα λατινικό μη υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Συμβιβαστική για γάμα μη. Ψήφισαν όλοι και όλες. Ε, απορρίπτεται 21-24. 124 υπέρ. Κατά. Yes. Εγκρίνεται. 120, 127 υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. εποχές εγκουρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα δέλτα λατινικονή υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Τώρα η 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 167 καταπίπτουν 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι υπόλοιπες κατά ύπτουν 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά Αποχές 143 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν 149 υπέρ κατά εποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά Yes. Απορρίπτεται 151 υπέρ κατά εποχές. Α, επαλήθευση απολύτευση. 151. Α, όχι, έχει ζητηθεί κατά τμήματα. ηλεκτρονικά όμως, ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 151. Τμήματα. Όχι, κατά τμήματα. Ψήφισαν όλοι υπέρ, ε, εντάξει. 40, 21 υπέρ, 23 σου κατά. Απορρίψτε. Απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά εποχές Γκρίνεται. 153 Πε, κατά εποχές εγκρίνεται 154 156 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γνωμοδότηση προϋπολογισμού 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ίδιο 5 Η επόμενη του προπολογισμού, λοιπόν, α, επαναλαμβάνει την προηγούμενη, ναι, έξι τώρα, η έξι του προπολογισμού, υπέρ, κατά, αποχές. Επαλήθευση για την παράγραφο 6 προϋ... γνωμοδότηση του προϋπολογισμού. Ναι. Τον προϋπολογισμό. Βίβησαν όλες. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7 υπέρ. Κατά. Yes. Ονομοδότηση Γνωμοδότηση απασχόλησης για την ενισχυμένη συνεργασία. Α, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε λοιπόν τότε. 162 υπέρ. Κατά. Χες. Γκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται προϋπολογισμός 1 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται προϋπολογία 3 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 5 υπέρ Κατά. παχες, Παλήθευση για την πέντε παρακαλώ. Εγκρίνεται 23-21. Η 6 και 7 καταπίπτουν 8 υπέρ. Κατά. παχες, Εγκρίνονται. Εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΙΕ όμικρον λατινικό υπέρ κατά χες επαλήθευση. Λήθευση. Ψήφισαν όλοι. δέκα υπέρ κατά χες εγκρίνεται. 11 καταπίπτει. 12 όμως, όχι, 12 υπέρ. Κατά, ποιες εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα την οικοπή υπέρ. Κατά, ποιες εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά, ποιες εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά, ποιες εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα ζήτα λατινικό Q υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται όπως οι άλλες, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Έληξε. Απορρίπτεται 21-23. 17 υπέρ. Κατά. Και επαλήθευση για τη 17. Επαλήθευση. Πάει αυτή. 22-23. 18 υπέρ κατά όχι εγκρίνεται 19 έχει καταπέσει 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα τα λατινικό ρο υπέρ, κατά, αποχές, Καραπορύπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι άλλες καταπίτουν 25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται είκοσι υπέρ κατά Δεν σηκώνετε το χέρι σας. Λοιπόν, επαλήθευση ηλεκτρονικά για την 27. 27. είναι ίδια με την 26, αλλά 26 έχει αποσυρθεί. Λοιπόν, εγκρίνεται η 27. 28 καταπίπτει, συμβιβαστική γιώτα θήτα, αλλά σίγμα υπέρ. Κατά εποχές. Εγκρίνεται συμβιβαστική κάπα, αλλά την έχει αποσυρθεί. 30 υπέρ κατά εγκρίνεται, οι υπόλοιπες καταπίπτουν, συμβιβαστική ΚΑΠΑ λατινικό Ι, έχει αποσυρθεί 33 και 34 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, η 35 έχει αποσυρθεί, η επόμενη συμβιβαστική έχει αποσυρθεί, 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μου φαίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 και 41 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 40 και 41. Εγκρίνεται η 42 εκπίστη συμβιβαστική ΚΓ λατινικό W, υπέρ, υπέρ, κατά, χες, απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 44 υπέρ α, α όχι παρασύρθηκα εδώ 47 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Χρωμοδότηση προϋπολογισμών Β υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Γ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονικά για το σύνολο όπως έχει τροποποιηθεί. Αμέσως κατευθείαν στο μηχάνημα. Κατευθείαν. Μετράω. Ψήφισαν όλες. Έληξε. Έληξε. Εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 14 αποχέ. Εγκρίνεται λοιπόν. Πάει. Εντάξει. 25 υπέρ τελικά. Ο κύριος Χάνς, Πέτερ και Μάρτιν. Εγώ θα είχα απόσχει, εάν είχα κάρτα, δεν έχω βέβαια. 15 αποχές επομένως. Κύριε Γκόκ, θέλετε να πείτε κάτι, ο εισηγητής. Δύο απλώς παρατηρήσεις. Ως εισηγητής για την έκθεση αυτή θέλω να εκφράσω τα αισθήματά μου, τα συναισθήματά μου καλύτερα. Όπως ξέρετε, με απογοητεύει το κείμενο πώς τροποποιήθηκε σήμερα. Ορισμένα στοιχεία ήταν αποτέλεσμα, ήταν αντικείμενο καλών συμβαστικών λύσεων Αλλά δεν έχουμε ακόμα βγει από την κρίση και μέσα στο πλαίσιο αυτό λυπάμαι που δεν καταφέραμε να έχουμε μια πιο φιλόδοξη και επιθετική συμβαστική λύση για να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να οδηγηθούμε σε μια ανάκαμψη. Γι' αυτό οι σύντροφοί μου και εγώ κρατήσαμε στάση αποχή στην τελική ψηφοφορία. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο που μας μένει μέχρι την Ολομέλεια για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε όλοι μαζί να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Well, um, thank you for that statement on behalf of... Καταγράφουμε την ε, δήλωση του εισηγητή. Κλείνει η ψηφοφορία, κλείνει η σημερινή συνεδρίαση. Καλό απόγευμα για σε όλους και όλες.